Τώρα, στη συνεδρίαση της 11ης Νοεμβρίου του 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημείωσε το αίτημα της Πάτσκης για την υπεράσπιση της κοινοβουλευτικής του ασυλίας σε σχέση με την διαδικασία ε, δικαστικής προσφυγής στα λιθουανικά δικαστήρια βάσει του κανόνα 6.3. Στα ο πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων ενημέρωσε τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι θα πρέπει το αίτημα αυτό να θεωρείται απαξιωθέν πλέον από τη στιγμή που έχει ψηφιστεί να, υπάρχει παρέκκληση από την Κοινοβουλευτική Ασυλία για το εν λόγω θέμα. Τα πρακτικά της συνεδρίασης θα υποβληθούν στο Κοινοβούλιο προς έγκριση στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης